Έχω μία ανακοίνωση. Μία τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης με βάση το άρθρο 140, παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού. Σύμφωνα και με, τις, με συνεννόηση με τις πολιτικές ομάδες, αύριο το, την Πέμπτη το απόγευμα η συζήτηση με βάση το άρθρο 122 για τους ε, κινδύνους που απορρέουν από την κατάσταση και τις εξελίξεις στην Αίγυπτο αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι, οπότε η προτινόμενη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης που είναι ακριβώς ε, η δήλωση της ΥΠΑ εκπροσώπου